θεωρούνται δεκτές το τελικό προσχέδιο της ημερήσιας διάταξης όπως έγινε δεκτό από τη διάσκεψη των Προέδρων την 5η 22 Σεπτεμβρίου του 2009 σας έχει ήδη διανεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 137 του κανονισμού. Με τη συμφωνία λοιπόν των πολιτικών ομάδων θα μου επιτρέψετε να σας προτείνω τις εξής αλλαγές για την ημέρα Τετάρτη σχετικά με τις προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες, η προφορική ερώτηση 001-08 του 2009 η οποία αναφέρεται ε, στη συγκεκριμένη οδηγία αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, η έκθεση της κυρίας Φαζόν για τον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι πολίτες θα πρέπει ή δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν λάβει θεώρηση για να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστίθεται με συζήτηση στην ημερήσια διάταξη αμέσως μετά τις παρεμβάσεις ενός λεπτού σήμερα το απόγευμα. Η τρίτη πρόταση αφορά τον τίτλο της δήλωσης της Επιτροπής για την πολιτική κατάσταση στις Ονδούρες στα πλαίσια του συζήτησης για τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2009 τροποποιείται δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Κατάσταση. Αύριο, την Πέμπτη, η πρόταση ψηφίσματος. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα για αύριο και θα δώσω το λόγο σε όποιον το επιθυμεί μετά. Η πρόταση ψηφίσματο της Ευρωπαϊκή τη Επιτροπή μάλλον Κοινωνικών Υποθέσεων για την ετήσια έκθεση Progress για το 2010, όπως επίσης και ο κατάλογος των δραστηριοτήτων, έγινε δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 88 του κανονισμού και εγγράφεται ε, στις, στην ώρα ψηφοφορίας αύριο. Ο κύριος Κασουλίδης έχει ζητήσει το λόγο. PP does not agree το ΕΛΚ δεν συμφωνεί με την αλλαγή του τίτλου ε, του σημείου της ημερησίας διατάξεως σχετικά με τις Ονδούρες. διότι στον τίτλο αναφερόμασταν στην 29η Νοεμβρίου, την ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών. Τώρα ζητείται η διαγραφή της ημερομηνίας μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη γενική συζήτηση και κρίνουμε ότι πρέπει να παραμείνει όσοι είχε ο τίτλος. Η διαδικασία προβλέπει στην περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσει σχετικά με τι προπάσεις τροποποίηση που συμφώνησαν οι πολιτικέ ομάδε να υπάρξει ψηφοφορία. Και γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να υπερασπιστεί την θέση την οποία εξέφρασε ο κύριος Κασουλίδης και κάποιος ο οποίος ε, να ε, μιλήσει κατά της άποψης αυτής και αμέσως μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Εφόσον υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν. Αλλιώς μπορούμε να ψηφίσουμε απευθείας. Ποια; Α, διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να διατηρηθεί η πρόταση αυτή η οποία έχει κατατεθεί γιατί είναι φανερό ότι έχουν καταρρεύσει οι διαπραγματεύσεις στην Ονδούρα. Η προτινόμενη εκλογή είναι πράγματι παράνομη και δεν έχει νομιμοποίηση τη στιγμή που ο Ασκόν, ο ήδη πρόεδρος της Ονδούρας, έχει ε, χάσει την εξουσία μετά από ένα πραξικόπημα. Εγώ λοιπόν ζητώ να διατηρηθεί η διατύπωση η οποία υπάρχει χωρίς να αναφέρεται στις εκλογές 29 Νοεμβρίου. Καλώς. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Ένας μόνο θα πάρει το λόγο. Ο κύριος Πέτερλε. Σας ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Πέτερλε. Okay. Jaz se zelo zavzemam za to, da ohranimo dnevni red nespremenjen. Jaz sem bil v delegaciji Evropske ljudske stranke, ki si je v Hondurasu imela priliko seznaniti z razmerami tam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 Ακούσαμε λοιπόν τις δύο απόψεις υπέρ και κατά της αρχικής πρότασης. Ας ψηφίσουμε παρακαλώ τώρα. Ψηφίζουμε λοιπόν για την τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης αποδεχόμενη τη φράση στα πλαίσια και των εκλογών που θα γίνουν στη χώρα αυτή. Ποιοι είναι υπέρ του να αφαιρεθεί το τμήμα αυτό που αναφέρεται στις εκλογές. Κατά. On, on your position, that, uh, okay. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ψηφίζουμε την πρόταση της Προεδρίας, η οποία ζητά την τροποποίηση του τίτλου, βάζοντας επιπλέον την μικρή φράση και τις εκλογές του 2009. Κατά. Νομίζω πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονική επαλήθευση. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό θέμα. Δεν έχω την, κάρτα μου γιατί δεν προβλεπόταν ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να καταγράψετε το ότι εγώ υπερψηφίζω την διατήρηση ημερήσιας διάταξης όπως είχε προταθεί. Δεν μπορεί ένα μηχάνημα να με αντικαταστήσει. Συνάδελφοι, πολλοί μπορεί να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Μην πάρετε το λόγο ο καθένας ξεχωριστά. μπορούμε να ακούσουμε την άποψή σας, μπορεί να περάσει η άποψή σας στα πρακτικά, αλλά δεν θα συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία η άποψή σας. Θα πρέπει να έχουμε πάντα την κάρτα μας, γιατί η αδίποτε στιγμή μπορεί να γίνει ψηφοφορία στην αίθουσα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Παρακαλώ, δεν θα γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα βάλουμε τις απόψεις σας στα πρακτικά. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της Προεδρίας. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 252 ψηφίσαντες, 109 υπέρ, 142 κατά. Μία αποχή. Η ημερήσια διάταξη παραμένει λοιπόν ως έχει. Allora, Πήγαμε πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα και διακόπτουμε τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής όπως προβλέπεται στη Μέση Διάταξη.